Το Πρώτο θέμα είναι η έκθεση που αφορά τη συμφωνία με την Ελβετική Συνομοσπονδία. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. εγκρίνεται το επόμενο θέμα έκθεση Σβόμποντα Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Νομική Προστασία των Υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Πέρας Εγκρίνεται επόμενη έκθεση περασε εγκρινεται επομενη Φερχόφστατ έχετε το λόγο Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί πρέπει να παρέμβω για το θέμα άρσης ασυλίας του κυρίου Σπάσκιτς. Ο κύριος Σπάσκιτς ε, πέστειλε μία επιστολή στον πρόεδρο Σούλτς ε, και θέλω να το στηρίξω, να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Και ο λόγος είναι ο εξής. Στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, άκουσαν δύο προτάσεις ε, που είπε ο κύριος Σουσπάσχιτς ε, για την δικαιοσύνη στην χώρα του. Εκτός πλαισίου, εκτός του υπολείπου λόγου του. Γιατί αυτό το οποίο είπε ήταν να μεταφέρει τα λόγια του Προέδρου της Λιθουανίας για την δικαιοσύνη στην χώρα. Σας ζητώ λοιπόν να το αναπέμψετε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για να ακούσει ολόκληρο τον λόγο του κυρίου Σπάσκετς η Επιτροπή και όχι μόνο τις δύο φράσεις που απέστειλαν οι αρχές της Λιθουανίας. Αυτό σας ζητάω μόνο. Μάλιστα έχουμε ένα αίτημα αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλει κάποιος να μιλήσει υπέρ. Υπέρ. Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Στην περίπτωση αυτή του ε, ασυλία του κυρίου Σπάσκιτ, ε, μιλήσατε για φράσεις. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ένας ευρωβουλευτής δεν μπορεί να τιμωρηθεί για δηλώσει τις οποίες δεν έκανε. Δεν έκανε. Αυτό είναι το νόημα τη Ασυλία. Μάλιστα, θέλει κάποιο να μιλήσει κατά. Ναι, κυρία Φρέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω εισηγήτρια αυτή τη έκθεση, οφείλω να υπογραμμίσω ότι ε, σε βάθο εξετάσαμε το θέμα στη Νομική Επιτροπή. Πρόκειται για μια συμπεριφορά ε, η οποία αφορά την ε, κοινοβουλευτική διαδικασία και τη κοινοβουλευτική δραστηριότητα ε, του κυρίου Ουσπάσκιτς ε, πρόκειται επομένως ε, για μια, ένα κακό προηγούμενο για το Κοινοβούλιο όσον αφορά την αίτηση της ασυλίας φερθήκαμε με τον τρόπο αυτό γιατί δεν υπήρξαν στοιχεία τα οποία να οδηγήσουν σε συμπέρασμα για Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ. Παρακαλώ διανατάσεως της χειρός. Κατά. Αποχές. Νομίζω να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. We vote on Ψηφίζουμε επί του αιτήματο του κυρίου Φερχόφστατ. Vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Ψηφίζουμε επομένως επί της εκθέσεως υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Η έκθεση της κυρίας Χαουτάλα, αίτηση άσεως βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Ζερόμ Λαβριγιώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση του κυρίου Χρυσόγονου Έτηση ε άρσεως βουλευτικής ασυλίας ε, του κυρίου Ζανούς Κόρβιν Μίκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα, η έκθεση του κυρίου Ντούντα σχετικά με την αίτηση άρσεως βουλευτικής ασυλίας ε, του κυρίου Θεόδωρου Ζαγοράκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενο αίτηση για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Επίσης, αίτηση για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις και προσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστοσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. έτηση για διαβούλευση με την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των δυνατοτήτων της Συνθήκης της Λισαβόνας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. έτηση για διαβούλευση με την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με πιθανές Εξελίξει και αναπροσαρμογέ των τροχουσών θεσμικών συνιστοσών τη ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενο θέμα. Η έκθεση της κυρίας Φανόη Χόιζεν. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και συμβάσεις. Συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε τις ε, ε, τροπολογίες ε, και θα δούμε ποιες χωριστές ψηφοφορίες έχουν ζητηθεί. Ψηφίζουμε επί του κειμένου, επί του συνόλου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, βεβαίως. Vote is closed. Adapted. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 16. Παρακαλώ. Ψηφίσαμε και ενώ ψηφίζαμε, εσείς κάνατε σχόλιο για την ψηφοφορία. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Επόμενο σημείο, η ε, ονομαστική ψηφοφορία για την ιδεολογική σκέψη 16, άρχεται. What is closed? Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 2, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 2, παράγραφος 2α. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, το ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρθό 13, παράγραφος 1, εισαγωγή σε δύο τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρθρο 13.1. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, διαγραφή του άρθρου 18, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία επί της προτάσεως της Κομισιόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. θα δώσω το λόγο ε, στην εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ζητήσω μια αναβολή της ε, ψηφοφορίας για αυτό το σχέδιο κανονισμού γιατί σύμφωνα με το 61.2 ε, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνει. Ωραία λοιπόν. Έχουμε ένα αίτημα αναβολή από την εισηγήτρια. Θα ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση Σίλβα Περέιρα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης Έχουμε εδώ την παράγραφο 6 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 σε δύο τμήματα. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν, με συγχωρείτε. 14, προτροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Σε δύο τμήματα χωριστά, στο πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28. Σε δύο τμήματα και πάλι χωριστά το πρώτο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 30 σε δύο τμήματα και πάλι. Για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Κατά. Αποχές. Η παλήθευση ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έχετε ψηφίσει όλη λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 38. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο ε, τμήμα προ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε λοιπόν το ολόκληρο το ψήφισμα, ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο. Συγχαρητήρια καταρχήν. Επόμενο σημείο είναι μια έκθεση, η έκθεση Πεντιτσίνη, ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη. Περνάμε στην πέμπτη παράγραφο, πρώτη τροπολογία υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, αρχικό κείμενο για την παράγραφο 6, σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Σηκώστε το χέρι σας παρακαλώ, κατά. Αποχές, Παλήθευση ηλεκτρονική. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παραγράφος 15 σημείο C και πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Σας παρακαλώ να υψώνετε το χέρι σας. Υπέρ, ώστε είστε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 18. Υπέρ. Έχει αποσυρθεί. Υπέρ. Και πάλι. Είμαστε στην 18. Υπέρ. Ψηφίζουμε υπέρ. Έχουμε λοιπόν ε, ονομαστική ψηφοφορία για την επαλήθευση εδώ στο σημείο αυτό. Υπέρ. Α, συγγνώμη, έχουμε την απόσυρση ενός αιτήματος για ονομαστική. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 47 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 48 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 σε τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση ηλεκτρονική. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Η, το, η δεύτερο, το δεύτερο τμήμα ε, καταπίπτει. Τρίτο λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63 παράγραφος σημείο π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 παράγραφος 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η παραγράφος 67, σημείο B, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική. εγκρίνεται. 67 σημείο C σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση ηλεκτρονική παρακαλώ. Λίγη η ηλεκτρονική ψηφοφορία εγκρίνεται. Παράγραφος 67, σημείο F σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται 71 υπέρ κατά άποχες επαλήθευση ηλεκτρονική λίγη απορρίπτεται παράγραφος 72 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, Ίσως λοιπόν να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 73. Σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος... Α, θέλετε να υπαλληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά. Πολύ καλά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 79. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Μετά την παράγουμε την τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, AB υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται στο εκτιμώντας AI υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Στο εκτιμώντας AAC υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Λίγη η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Λοιπόν, το ψήφισμα ολόκληρο, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Uh, Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση DeBacker Ευκαιρίες Πράσινης Ανάπτυξης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παράγραφος 7 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 11 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 15 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Μέρος τρίτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή παράγραφος 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή παράγραφος 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε Πέρας. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Παράγραφος 32, υπότιτλος ονομαστική ψηφοφορία έρχεται». Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33 σε τρία μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 34 σε τρία μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται μέρος δεύτερο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Μέρος τρίτο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 35 σε 4 μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε πέρας Εγκρίνεται. Μέρος τέταρτο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παραγραφός 36 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 37 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 39 σε δύο μέρη. Υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 42 να την επαληθεύσουμε να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος πέρας απορρίπτεται Παράγραφο 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας γάμα σε δύο μέρη υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας ε, ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας κάπα σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας L σε τρία μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας. Τελειώσαμε. Ήταν και η πρώτη ψηφοφορία στην οποία προέδρευσα. Την ε, άδελφη. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτη έκθεση, έκθεση Χάιζεν. Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως μέσα σε χρηματοοικονομικά μέσα και συμβάσεις. I give the floor, uh, um, Mrs. Gill. Η κυρία Γκίλ έχει το λόγο. Um, thank you. Σας ευχαριστώ.